Λοιπόν, κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης που είχε αρθεί την προηγούμενη φορά στο Στρασβούργο. Τα πρακτικά της προηγούμενης συνόδου υπάρχουν στους φακέλους σας. Μήπως υπάρχει κανένα σχόλιο επ' αυτόν η παρατήρηση, όχι, εγκρίνονται. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Την Δευτέρα επλήγει η Ουγγαρία από τη χειρότερη θεομηνία της ιστορίας της. Δηλαδή τοξικά υγρά διέφυγαν από μία αποθήκη. Υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες. Θα ήθελα λοιπόν να στείλουμε τηλεγραφήματα συλληπιτήρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα τώρα να σας πω ότι αύριο θα γιορτάσουμε, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι, την τέταρτη επέτειο της δολοφονίας της Άννας Πολιτικόσκαγια που όπως ξέρετε είχε δώσει τη ζωή της για να ανακαλύψει την αλήθεια για αυτά που συνέβαιναν στον Κάφκασο στην Τσετσενία. Έχουμε ήδη αποτίσει φόρο τιμή στη μνήμη της κυρίας Πολιτικόφσκα για στον αγώνα της για την ελευθεροτυπία και την ελευθερία της έκφρασης αφού δώσαμε το όνομά της σε μία από τις αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά δεν ξεχνούμε ούτε άλλους δολοφονηθέντες δημοσιογράφους, την κυρία Αναταλία Εστεμίροβα και την κυρία Αναστασία Μαρμούροβα καθώς και άλλους αγωνιστές νομομαθείς όπως τον κύριο Στανισλάβ Μαρκελόφ, Σεργέη Μανίτκι και άλλους. Οι συνθήκες της δολοφονίας τους δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί και ζητούμε από τις ρωσικές αρχές να κάνουν ό,τι μπορούν για να σεβαστούν τις αρχές του κράτους δικαίου και να θερματίσουν επιτέλους αυτή την κατάσταση αβεβαιότητας. Στις 10 Οκτωβρίου θα εορτάσουμε την Διεθνή ημέρα κατάργησης θανατικής ποινής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να οργανώσει όπου μπορεί σε όλες τις χώρες ένα μορατόριο κατά της θανατικής ποινής. Δεν μπορεί να θεωρηθεί η θανάτωση ως καταδίκη νόμιμη βλέπουμε ότι και στη Ρωσία, στον Μπουρούντι και στο Τονγκό γίνονται κινήσεις για την κατάργησή της. Δυστυχώς όμως στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Ιαπωνία εφαρμόζονται ακόμη θανατικές εκτελέσεις. Φρονούμε ότι η δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, αλλά αυτό που μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι ο αριθμός των εκτελέσεων που συμβαίνουν σε χώρες όπως η Κίνα ή το Ιράν ζητούμε από τις αρχές των χωρών αυτών να τερματίσουν την πρακτική αυτή. Κυρίες και κύριοι, έλαβα από την ομάδα του ΕΛΚ αιτήματα ορισμού μελών ορισμένων αντιπροσωπείων Εάν δεν ακουστούν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα εγκριθούν οι ορισμοί αυτοί. Και τώρα κυρίες και κύριοι περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Σήμερα και αύριο, με σύμφωνη γνώμη των πολιτικών ομάδων, θα προτείνω τις εξής αλλαγές. Οι περισσότερες πολιτικές ομάδες είναι υπέρ των αλλαγών αυτών. Λοιπόν, ειδού την Τετάρτη, σήμερα δηλαδή, θα προσθεθεί στην μέση διάταξη ένα νέο σημείο η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τις κοινωνικές ρήτρε της ε, συνθήκης της Λισαβόνας μετά από, μετά από τη συζήτηση για τη βιοπικιλότητα. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε για την διαγραφή της προφορικής ερώτησης για τα εμπορευματοκιβώτια που χάνονται στη θάλασσα και την Πέμπτη να αρχίσουν οι ψηφοφορίες στις 11.30 αντί στις 11.00 και την Πέμπτη επίσης να διαγραφεί η συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Μάνικα ως προς τον διορθωτικό προπολογισμό 2-2010 διότι το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει και επομένως δεν υπάρχει λόγος να γίνει η συζήτηση αυτή αύριο. Τώρα, ως προς αυτό που σας είπα για σήμερα, για τα εμπορευματοκιβώτια, μπορείτε αν θέλετε να σχολιάσετε. Ο κύριος Βόρτμαν Κόλ έχει ήδη ζητήσει το λόγο. Η κυρία. κυρία. Κύριε Πρόεδρε, το ΕΛΚ πάντοτε δέχεται συζήτηση για κοινωνικά θέματα στις Ολομέλειες. Πρέπει όμως οι συζητήσεις αυτές να είναι σωστά προετοιμασμένες και γι' αυτόν τον λόγο στη διάσκεψη των Προέδρων